Okay, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, let's start our uh, session for today. Uh, We start with uh, agenda point 14. It's a... Καλημέρα. Καλημέρα. Προχωράμε στο σημείο 14 που είναι η παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Σλοβακικής Προεδρίας. Χαιρόμαστε που έχουμε μαζί μας τον κύριο Πίτερ Ζήκα που είναι ο Υπουργό Οικονομίας της Σλοβακίας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην Επιτροπή μας, την ΙΝΤΕ, εδώ στις Βρυξέλλες. Όλοι θα γνωρίζετε τις μεγάλες προκλήσεις, τις εμπορικές που θα έχουμε μπροστά μας. Θα τα συζητήσουμε αυτά, θα συζητήσουμε την συμφωνία ΣΕΤΑ βέβαια, για τις πρώτες υπογραφές, το θέμα των εξαιρέσεων στις προσωρινές ε, διατάξεις. Είναι ένα θέμα που συζητείται ευρέω. Ένα άλλο ζήτημα που θα μας απασχολήσει, που είναι επίσης σημαντικό για την οικονομία και τη βιομηχανία, είναι το θέμα του εξυγχρονισμού των ε, τρόπων που έχουμε να προχωρήσουμε σε εμπορικές διευθετήσεις και διατησίες. Θα έχουμε περισσότερα νέα το Δεκέμβριο. Θα δούμε λοιπόν πώς θα βρούμε το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε και καλές λύσεις. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μαζί πρέπει να έχουν αποφασίσει πριν από την 10η Δεκεμβρίου. Υπάρχουν και νομοθετικά ζητήματα, νομοθετικοί φάκελοι. Όσον αφορά τα ορυκτά, είναι ένα. Ένα άλλο είναι διαπραγματεύσεις που θα αρχίσουν με την Ιαπωνία. Μπορεί να προχωρήσει αυτό το θέμα. Και βεβαίως Έχουμε και την πολυμερή προσέγγιση και την πρόοδο στην Γενέβη. Πολλά έχετε μπροστά σας. Ενδιαφέροντες καιροί. Οπότε είμαστε πολύ περίεργοι να σας ακούσουμε, να μας εξηγήσετε πώς θα τα αντιμετωπίσετε όλα αυτά. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας, κύριε Λάγκερ. Κυρίες και κύριοι, είναι χαρά που βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και που έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας πολύ σημαντικά ζητήματα όπως είναι το εμπόριο και η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προνόμιο για μένα και συγχρόνως βέβαια και πρόκληση για την Σλοβακία που αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης. Θέλω σε αυτήν την συνάντηση να σας παρουσιάσω τις προτερότητές μας για τους επόμενους έξι μήνες όσον αφορά το εμπόριο και την εμπορική πολιτική. Πρώτον, θέλω να σας πω ότι εκτιμώ όλους ιδιαίτερο το σκληρό έργο των προκατόχων μας και του τρίου. Έτσι έχουμε μια στέρεα βάση πάνω στην οποία να προχωρήσουμε και εμείς και να συνεχίσουμε με καλό πνεύμα συνεργασίας με όλες τις χώρες μέλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Σλοβακία είναι ανοιχτή χώρα, προσανατολισμένη στο εμπόριο, στις εξαγωγές και βλέπει ότι υπάρχουν θετικά πλεονεκτήματα από τα οποία υποφελείται η ανάπτυξη και η απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα η επενδυτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μεγάλη σημασία και μαζί με τις χώρες μέλη, την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Σλοβακική Προεδρία θέλει να βοηθήσει προκειμένου να πετύχουμε πραγματικά ωφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες και την οικονομία των χωρών μας. Θέλω επίσης να υπογραμμίσω το θέμα της διαφάνειας, της ενημέρωσης, που βοηθάει σε αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των πλευρών. Τώρα, θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου όσον αφορά την εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προτεραιότητές μας. πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες έγκρισης για να προετοιμαστούμε για την υπογραφή της ε, συνολικής ε, συμφωνίας ΣΥΤΑ με τον Καναδά. Διαπραγματεύσεις επίσης όσον αφορά το TTIP θα είναι οι κύριες προτεραιότητε της Προεδρίας μας. Όσον αφορά την ε, σημερινή κατάσταση της Ευρωπαϊκής Καλλιβουργίας, τον ανταγωνισμό, την προστασία σημάτων, αντιμετώπιση dumping, υπάρχει πρόταση για τον εξυγχρονισμό του σημερινού ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου. Η Προεδρία μας λοιπόν έχει ακούσει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και προσπαθεί να πετύχει πρόοδο στον εξυγχρονισμό αυτό ακούγοντας όλες τις πολιτικές απόψεις, και όσον αφορά το θέμα του καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα, την απόδοση του καθεστώτος αυτού δηλαδή. Σίγουρα όλα αυτά αποτελούν πολύ σημαντικές προκλήσεις για την Προεδρία μας. Τέλος, αλλά και λιγότερο σημαντικό, δεν πρέπει να ξεχνάμε και το, την πολυεπίπεδη προσέγγιση. Πρέπει να δούμε τη θέση μας στον ΠΟΕ, που είναι και ο θεματοφύλακας των πολυμερών εμπορικών συστημάτων. Με την αυτή προεδρία, λοιπόν, θέλουμε να αποτελέσουμε έναν επικοδομητικό εταίρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εμπορική και επενδυτική στρατηγική μας και να συμμετέχουμε σε όλες τις διαδικασίες διαπραγματεύσεων Πάντως, θα προσπαθούμε να προσαρμοζόμαστε και στις νέες εξελίξεις ε, μετά τα πρόσφατα νέα που έχουμε από τον Ηνωμένο Βασίλειο. Τις επόμενες μέρες και μήνες θα προχωρήσουμε με την πολιτική μας, πάντως βάσει του άρθρου 50 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ενεργοποιήσει το άρθρο αυτό 50, παραμένει πλήρες μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα. Θα δούμε τι θα γίνει εφόσον υπάρξουν ε, διαπραγματεύσεις, πώς θα προχωρήσουν αυτές, εφόσον μία από τις πιο σημαντικές μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί πλέον μέρος της. Τώρα, υπογραφή της ΣΕΤΑ, της συμφωνίας με τον Καναδά δηλαδή αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για την Προεδρία. Είναι μια πολύ καλή συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνεισφέρει στην ενίσχυση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Γι' αυτό και πρέπει να υποφεληθούμε όσο γίνεται πιο γρήγορα από τα ωφέλη που μας προσφέρει. Τώρα που η Επιτροπή έχει υποβάλει στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πρόταση της για υπογραφή, έχει αρχίσει το έργο στο Συμβούλιο για να Υπογραφή στις 27 Οκτωβρίου η συμφωνία αυτή στη διάσκεψη κορυφής Ευρωπαϊκή Ένωσης Καναδά. Ήδη από το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε πει ότι πρόκειται για μια μεικτή συμφωνία και ότι έτσι θα την διαπραγματευόταν. Έχει υποβληθεί λοιπόν η συμφωνία ως τέτοια στο Συμβούλιο. Η κύρωση πρέπει να περιλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και είναι μεικτή συμφωνία αυτή, όπως έχουν ζητήσει και τα διάφορα κοινοβούλια, αλλά και η κοινή γνώμη. Μετά την υπογραφή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ζητηθεί να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του. Το Φεβρουάριο του 2016 ανακοινώθηκε το πέρασμα στην τελική διαδικασία με μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την προστασία σε περίπτωση διενέξεων. με τους επενδυτές. Έτσι έχουμε προχωρήσει σε ένα νέο μοντέλο για την ε, προστασία των επενδυτών και για την ε, διαδικασία διαιτησίας. Συνεχίζουμε και με τις την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας που είναι πολύ βασικό για την αξιοπιστία μας απέναντι στον Καναδά. Είναι βέβαια πολύ νωρίς να προκαταλάβουμε τι θα βγει από τις συζητήσεις. Πάντως οι διατάξει όσον αφορά τις επενδύσεις απαιτεί ένα νέο σύστημα το οποίο δεν θα εφαρμοστεί ακόμα. Για το TTIP τώρα. Και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία πριν από τα τέλη της χρονιάς αυτής. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδο τους τελευταίους μήνες, όμως παρόλα αυτά παραμένει πολύ σκληρή δουλειά. Ο επόμενος γύρος θα είναι πολύ σημαντικός για την επιτυχία. Αγωνιζόμαστε πάντως για να έχουμε υψηλέ φιλοδοξίες και από τις δύο πλευρές. Δεν θα συμφωνήσουμε ε, για τη συμφωνία αυτή απλώς και μόνο για να έχουμε μια συμφωνία. Όχι, θέλουμε υψηλέ προδιαγραφές γιατί αυτός είναι ο μόνος σωστός τρόπος. Δεν μπορούμε να έχουμε όμως ούτε ένα TTIP light. Θέλουμε από τη συμφωνία αυτή να υποφεληθεί ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρε ε, μέλη σε όλου του πυλώνε, είτε πρόκειται για την πρόσβαση στην αγορά, είτε πρόκειται για τι υπηρεσίε, είτε πρόκειται για τι δημόσιε συμβάσει, τα μη δεσμολογικά μέτρα κλπ. κλπ. Η διαπραγματευτική εντολή τηρείται. Προσπαθούμε να μην πέσουν καθόλου οι προδιαγραφές στα στάνταρτς των χωρών μελών και να μην υπάρξει ελευθέρωση για το εκπαίδευση, υπηρεσίες. Όσον αφορά τώρα την προστασία των επενδυτών, η Ευρωπαϊκή Ένωση πιέζει για ένα νέο μοντέλο με ένα νέο σύστημα δικαστικό που να ρυθμίζει τέτοιου είδους διενέξεις. Οι υπουργοί την επόμενη φορά που θα συναντηθούν θα σημειώσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και θα καθορίσουν το δρόμο για τη συνέχεια. Τώρα όσον αφορά για την πρόσβαση των Ευρωβουλευτών αλλά και των Εθνικών Βουλευτών στα έγγραφα διαπραγματεύσεων, προσπαθούμε να πετύχουμε τη διαφάνεια και να διασφαλίσουμε δημοκρατικό έλεγχο. Όμως έχει υπάρξει διαρροή των εγγράφων από την TTIP, κάτι το οποίο δεν είναι προς όφελος κανενός. Γιατί έτσι υπονομεύεται η αξιοπιστία, η διαπραγματευτική μας θέση, και η πρόσβαση σε επόμενου είδους διαπραγμάτευση. Ελεύθερο εμπόριο με την Ιαπωνία. Υπάρχει πρόοδος όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία αυτή, αλλά δυστυχώς πάμε πάρα πολύ αργά, απογοητευτικά αργά. Θα θέλαμε να ολοκληρώσουμε στο, μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργό το Μάιο που μας πέρασε. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει να επιταχυνθεί ο ρυθμός, να υπάρξει πολιτική συμφωνία, κυρίως από πλευράς της Ιαπωνίας, για να αντιμετωπιστούν τα πιο δύσκολα και σε κρεμότητα ζητήματα. Ο στόχος για την Προεδρία μας είναι να συνεχίσουμε να μικραίνουμε το χάσμα, τις διαφορές δηλαδή που παραμένουν μεταξύ μας. Επιπλέον, από το ΣΕΤΑ, ΤΙΤΙΠ και η Ιαπωνία, έχουμε διαπραγματεύσεις και με άλλους εμπορικούς εταίρους. Θα σας αναφέρω μερικούς από αυτούς. Μερκοσούρ. Δίνουμε μεγάλη σημασία στα συμπεράσματα της συνολικής μας συμφωνίας με το Μερκοσούρ που έχει να κάνει με τα συμφέροντα μετικά και άλλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο θέμα των αγαθών, των δημοσίων ε, συμβάσεων, υπηρεσιών και θέλουμε να ξαναμπούν διαπραγματεύσεις στις ράγες. Υπάρχει και το θέμα του νερού που μας απασχολεί για τη Γεωργία. Και το πιο, το πιο ευαίσθητα προϊόντα το βιοκρέας για παράδειγμα έχει αποκλειστεί και το μοσχαρίσιο κρέας. Υπάρχουν προκλήσεις πολλές για τη Γεωργία. Περιμένουμε τις τελικές ε, αποφάσεις και να μελετήσουμε και τον ε, αντίκτυπο συμφωνιών όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Γεωργία μέχρι το Σεπτέμβριο. Εκουαδόρ. σήμερινο για Κολομβία, Περού επίσης. Όσον αφορά την εφαρμογή ενός πρωτοκόλου προσχώρηση σε τέτοια συμφωνία πριν από τα τέλη του 2016 με εμπορικά ε, μέτρα, επειδή η προηγούμενη συμφωνία με το Εκουαδόρ εκπνέει. Μας πήρε δύο χρόνια μετά τις διαπραγματεύσεις με τον Ισημερινό για να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει. Το Συμβούλιο κάνει ό,τι μπορεί για να υπογραφεί η συμφωνία τον αύριο. Περιτώ να πω ότι τόσο ο σημερινός όσο και η Κολομβία και το Περού πρέπει να είναι έτοιμες για να μην υπάρξουν παρετέρω καθυστερήσεις. Είμαστε σίγουροι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναλάβει το ρόλο του και θα φροντίσει έγκαιρα να ολοκληρωθεί η διαδικασία, ώστε το, ο σημερινός να πάρει την υποστήριξη που χρειάζεται σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει. Η Σλοβακική Δημοκρατία χαίρεται που μπορούν να αρχίσουν και διαπραγματεύσεις με το Μεξικό μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Οι πρώτες επίσημες διαπραγματεύσεις θα λάβουν χώρα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Υπάρχουν πολλές φιλοδοξίες για τον εξυγχρονισμό του εμπορίου σε μια συνολική συμφωνία και με ένα δεσμευτικό πλαίσιο όσον αφορά τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Μεξικό. Επιτρέψτε μου τώρα να στραφώ σε διάφορους νομοθετικούς φακέλους που θα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Την απόδοση του καθεστώτος της οικονομίας της αγοράς στην Κίνα. Είναι χωρίς προηγούμενο σημασίας πολιτικό στίγμα που θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τεράστιες επιπτώσεις διότι θα επηρεάσει όχι μόνο το ευρωπαϊκό εμπόριο, αλλά και την απασχόληση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της στα πλαίσια του ΠΟΕ και πρέπει να προσαρμόσει και την ομοθεσία της που έχει να κάνει με τους παραγωγούς ώστε να έχει εμπορικό εταίρο την Κίνα. Η πρόταση υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα το Συμβούλιο για την απόδοση του καθεστώτος αυτού στην Κίνα, αλλά ούτε και για προϋποθέσεις προκειμένου να βληθούν μέτρα ώστε να μπορέσει να γίνει εφικτή μια τέτοια απόφαση. Προσβλέπουμε λοιπόν στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και την Επιτροπή, δηλαδή και τα τρία θεσμικά όργανα, προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Εξετάζουμε πάντως τις επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια απόφαση. Το Συμβούλιο έχει κάνει προπαρασκευαστικό έργο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δημόσια διαβούλευση με όλες τις πλευρές. Στα πλαίσια τώρα της σημερινή κρίσης στην Ευρωπαϊκή Χαλιβουργία έχει αρχίσει τεχνικές συζητήσεις στο Συμβούλιο για τις 20 προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τον εξυγχρονισμό των ε, εμπορικών αμυντικών μέσων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να δούμε πώς θα βελτιώσουμε τους μηχανισμούς μας αυτούς, να προσαρμόσουμε τις εμπορικές μας πρακτικές για να ενισχυθεί η ανταγωνιστική μας θέση και οι ευρωπαϊκές ε, επιχειρήσεις να μην βρίσκονται σε κατώτερη μοίρα από άλλες. Λαμβάνουμε υπόψη δυνατότητες επιτάχυσης των διαδικασιών για παράδειγμα και εξετάσουμε και την αλλαγή της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των περιθωρίων κέρδους. Είναι θετικό το Συμβούλιο για πολλές από τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρ' όλα αυτά είναι διχασμένες οι απόψεις στο Συμβούλιο, κυρίως για τη μερική εφαρμογή του lesser utility. Νομίζω ότι σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι βέβαια πολύ νωρί να πούμε ποιε από τις ιδέες που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα γίνουν αποδεκτές τελικά από τις χώρες μέλη και ποιε όχι. Ω Προεδρία θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διευκολύνουμε ένα σεβιβασμό στο Συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσουμε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο γίνεται πιο γρήγορα για την τελική απόφαση. Διεθνείς συμβάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αντιμετωπίσει κάποιε ανισορροπίε που υπάρχουν μέχρι τώρα όσον αφορά την πρόσβαση στι δημόσιε συμβάσει στι αγορέ τρίτων χωρών. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η πρόταση του IPI θα είναι ισορροπημένη, ότι δεν θα αυξήσει το διοικητικό άκθο τη γραφειοκρατία και δεν θα στρεβλώνει την ανταγωνιστικότητα της εσωτερικής μας αγοράς. Ούτε θα υπάρχουν και αρνητικέ αντιδράσεις, αντίπεινα ουσιαστικά από τρίτες χώρες. Πρέπει να πω ότι η κατάσταση στο Συμβούλιο είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και ακούγονται διαφορετικές απόψεις από τις χώρες μέλη. ΠΟΕ. Εμπορικές πολιτικές και διαπραγματεύσεις για περιφερειακές συμφωνίες. Υπάρχει εδώ το θέμα της πολυεπίπεδης προσέγγισης. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τον ΠΟΕ γιατί πιστεύουμε ότι αποτελεί θεματοφύλακα τέτοιων πολυεπίπεδων εμπορικών συστημάτων. Δουλεύουμε για την εφαρμογή των συμπερασμάτων της Υπουργικής διάσκευσης του ΠΟΕ, που είναι για το μετά τον Αιρόμπι πρόγραμμα, όπως λέγεται και αφορά συμφωνίες πολυεπίπεδες σε υπηρεσίες, ε, περιβάλλον κλπ. Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, τελειώνοντας θέλω να υπογραμμίσω ότι η διαφάνεια, η πρόσβαση στην ενημέρωση, αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων είναι ζωτική σημασία. Πολλά διακυδεύονται εδώ, σημαντικά, αλλά εμεί θα δραστηριοποιηθούμε, θα φροντίσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί, να αποδώσουμε έργο για να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του εμπορίου με ρεαλιστικέ φιλοδοξίε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και προσβλέπω τώρα σε συζήτηση μεταξύ μα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ε, θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και μετά στα άλλη μέλη. Και να ξέρετε ότι έχουμε μισή ώρα στη διάθεσή μας. Γιατί μέσα σε αυτή τη μισή ώρα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον Υπουργό και να απαντήσει. Προτείνω λοιπόν ο κάθε ένας από εσάς ε, να μιλήσει για δύο περίπου λεπτά το ΕΛΚ, η πρώτη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα, ο κύριος Βίνκλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά που μας ε, είπατε που ήταν πραγματικά μια πολύ εκτεταμένη και ευρία προσέγγιση. Δεν ξέρω αν θα σας φτάσουν ε, οι έξι μήνες για όλα αυτά, ίσως χρειαστείτε περισσότερο χρόνο. Βάση περιπτώσει, εγώ σας συγχαίρω για την προσέγγιση σας. Επειδή ξεκινήσατε με τη συμφωνία ΣΥΤΑ, θα ξεκινήσω και εγώ με αυτή τη συμφωνία, η οποία είναι πολύ σημαντική για το ΕΛΚ. Υπάρχει ο ακρογωνιαίος ε, λίθος ε, που είναι αυτή η συμφωνία. Η επικύρωση από τα Εθνικά Κοινοβούλια είναι πολύ σημαντική, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλές ε, διαπραγματεύσεις που έπονται, ε, υπάρχουν οι προσδοκίες των επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων ε, και από τις δύο πλευρές, τόσο δηλαδή από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από τον Καναδά. Πράγματι αυτή η συμφωνία μπορεί να στηρίξει τις οικονομίες μας, την αναζήτηση θέσεων απασχόλησης ε, και αυτό το θέμα θα συζητηθεί το φθινόπωρο στη συνάντηση κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση Καναδά. Πάντω, η προσωρινή εφαρμογή είναι πολύ σημαντική. Πρέπει λοιπόν να υπογράψουμε σε αυτή την συνάντηση κορυφή, να αρχίσει να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω ότι ε, κατά πόσον το 90 κάτι ε, τη συμφωνία είτε αφορά το εμπόριο. Πάντως το μεγαλύτερο ε, ποσοστό της συμφωνίας αφορά πράγματι τις εμπορικές ανταλλαγές. Μιλήσατε για την αξιοπιστία και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα, αλλά ακόμα πιο σημαντικό είναι το ενδιαφέρον των εταιριών μας ε, και τα συμφέροντα των, της οικονομίας μας. Η θέση της, της Κίνας Πράγματι, εχθές διαβάσαμε τις δηλώσεις ε, στη συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Διαβάσαμε αυτά που είπε ο κύριος Γιούγκερ, που είπε ότι η οικονομία της αγοράς ε, και οι προπολικέ δυνατότητε που προσφέρει η Κίνα, αυτά τα δύο είναι άρρηκτα συνδεμένα μεταξύ τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει λιγάκι να περιμένουμε ακόμα, περιμένουμε ακόμα τις δηλώσεις της Επιτροπής ε, για συγκεκριμένα θέματα. Τα ορυκτά. Πράγματι, πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχει η προσέγγιση της ε, Τρόικα, υπάρχει η κληρονομιά από την ε, Ολλανδική Προεδρία. Παρακολουθούμε να ακολουθήσει αυτή την κατεύθυνση. Εκ μέρου των ε, Σοσιαλδημοκρατών, Ροντρίγκε, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σα ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ σήμερα. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε κάποια ζητήματα θέλω κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις. Αναφερθήκατε στην σημασία της διαφάνειας, ένα βασικό στοιχείο για το Κοινοβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω πώς αξιολογείτε τις εντολές για τη διαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών. Για την Τινησία, ας πούμε, δεν ξέρω ακόμα το περιεχόμενο της εντολής. Δεν θεωρείτε ότι άμεσα θα πρέπει το περιεχόμενο της εντολής να δημοσιοποιηθεί. Για την αντίστοιχη ξέρετε ότι έχουμε διαφορές μεταξύ του Κοινοβουλίου που εξέφραστε σε αυτή με ευρία πλειοψηφία και τη θέση που εκφράζει η Κομισιόν. Ποια είναι η θέση σας από αυτού. Όλες οι εμπορικέ συμφωνίες θα πρέπει να γνωρίζετε ότι εγκρίνονται εδώ στο Κοινοβούλιο, οπότε είναι απαραίτητο να εισακούονται οι συστάσεις μας για το Μερκοσούρ. Θέλω τη γνώμη σας για την μη περιλήψη ενός κεφαλαίου. Ίσως αυτή η παράληψη να έχει κάποιο λόγο παλαιότερα. Αλλά σήμερα δεν νομίζω να υπάρχουν ακόμα λόγοι για να μην υπάρχει αυτό το κεφάλαιο για την προστασία των επενδύσεων. Για την Νότιο Αμερική λυπάμαι που δεν αναφέρατε την Χιλή. Χιλή η οποία έχει ξεκινήσει μία διαδικασία εξυγχρονισμού και η κυρία Μάστρομ και η κυρία Μογκερίνη έχουν αναφερθεί αλλά δεν αναφέρθηκε από εσά στην αρχική σας ομιλία. Θα ήθελα να μου πείτε λοιπόν υπό την Προεδρία σας τι θα κάνετε με το θέμα της Χίλης. Ευχαριστώ. E Ευχαριστώ, Τσαχαντήλ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας πω ότι χαίρομαι που η Προεδρία μετακινήθηκε επιτελούς στην γειτονιά μας στην Κεντρική Ευρώπη. Η χώρα μου έχει πολιτική ιστορία, κοινή ιστορία με τη Σλοβακία. Πάντως εγώ άκουσα με ενδιαφέρον αυτά που είπατε και μου επιβεβαίωσαν αυτό που περίμενα. Δηλαδή ότι η Σλοβακία είναι μια χώρα εξαγωγική και ανοιχτή. Ο Υπουργός μας παρουσίασε όλες τις πολυμερείς και διμερείς σημαντικές συμφωνίες. Μας μίλησε για τις υποεξέλιξη διαπραγματεύσεις. Το έκανε με τρόπο νομίζω αρκετά επαγγελματικό. Και βεβαίως στη συνέχεια Θα ακούσουμε στο τέλος μια περιγραφή της περίπλοκης σχέσης που υπάρχει. Εννοώ με αυτό την απόδοση του καθεστώτος οικονομίας αγοράς στην Κίνα. Βέβαια ταυτόχρονα θα πρέπει να προστατεύσουμε και τις ντόπιε της εχώριες παραγωγές μας, ιδιαίτερα εκεί όπου είναι ισχυρές, όπως ας πούμε τη χαλιβουργία. Χάρηκα λοιπόν που το αναφέρατε αυτό. Δεν έχω στην ουσία ερωτήσεις. Θα να σας πω κυρίως ότι σύμφωνα απόλυτα και χαίρομαι για το σχέδιο της Σλοβακικής Προεδρίας και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ελπίζω να πετύχετε όλους τους στόχους που έχετε θέσει και είμαι βεβαίως ότι η Επιτροπή μας εδώ θα είναι πάντοτε στο πλευρό σας και θα σας στηρίξει. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για όλα αυτά που μας είπατε. Όπως ίσως θα έχετε ακούσει, κάποιοι διαδηλωτές ε, έχουν μπλοκάρει ένα κομμάτι της πόλης γιατί σήμερα γίνονται διαπραγματεύσεις για το TTIP και το σύνθημά τους ε, είναι ότι πάει τέλειωσε το TTIP, τέλος με το TTIP. Αυτό δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι. Game over λένε συγκεκριμένα στα αγγλικά. Εσείς τι πιστεύετε, ποια είναι η δική σας άποψη, γιατί μας παρουσιάσετε εδώ μια πολύ φιλόδοξη ένα πολύ φιλόδοξο θεματολόγιο και ένα βασικό θέμα είναι τι θα γίνει στη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Καναδά και ε, επίση να έχετε κατά νου το τι θα προκύψει εάν αποτύχει αυτή η διαδικασία επικύρωσης. Ήθελα επίση να σας ζητήσω να μας εξηγήσετε λιγάκι το τι ακριβώ εννοείται με την ε, προσωρινή εφαρμογή τη συμφωνία ΣΥΤΑ. Αν κατάλαβα καλά, εσείς θέλετε προσωρινά να εφαρμοστεί το κομμάτι που αφορά στις ε, επενδύσεις και στη βιομηχανία. Αυτή είναι η θέση του Συμβουλίου ή μήπως είναι η ποιος ειναι η θεση της κυβέρνησής σας. Και επίση, μήπω μπορείτε να μα ενημερώσετε λιγάκι το πώ ερμηνεύει το Συμβούλιο αυτέ τι συμφωνίε. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απομακρύνεται από τι συμβουλέ τη Ενωμική Υπηρεσία ε, για πολιτικού λόγου. Ε, Βεβαίω το Συμβούλιο και όπω πολύ καλά γνωρίζετε οι Υπουργοί δεν χρειάζονται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απευθυνθούν στα εθνικά του κοινοβούλια, για να ψηφίσουν αυτά έτσι τα εθνικά κοινοβούλια να συμμετάσχουν στις συζητήσεις ευθύς εξ αρχής σε όλα αυτά ε, που διαδραματίζονται λόγω των συμφωνιών. Μπορούν να αρχίσουν αυτά να εφαρμόζονται ε, στην περιφέρεια, στην τοπική κοινωνία, από την κοινωνία των πολιτών, παντού. Άρα δηλαδή ε, εδώ έχουμε μια πολύ σκληρή δοκιμασία για την ΣΥΤΑ και σας ερωτώ, εσείς τελικά αν τελειώσει, κλείσει το θέμα της ε, ΣΥΤΑ. Ε, Ποιε θα είναι οι συνέπειες, θα υπάρχουν συνέπειες ε, στις διαπραγματεύσεις όπου ίσως οι χώρες αρχίσουν πάλι να ανταγωνίζονται μία την άλλη σε παγκόσμιο επίπεδο. Και τέλος, κάποιες παρατηρήσεις που είπατε για τη διαφάνεια. Γιατί το Συμβούλιο δεν δημοσιεύει τις εντολές που δίνει ε, στο πλαίσιο των εμπορικών διαπραγματεύσεων, όπως αυτή για την, την Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο πιέζουμε για την ε, διαφάνεια, τη χρειαζόμαστε απαραίτητο την ε, διαφάνεια και τελικά από ό,τι φαίνεται το Συμβούλιο είναι εκείνο το οποίο διαφωνεί με τη δημοσίευση των εντολών. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα για την Γκουε, επόμενος ομιλητής, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και τον κύριο Υπουργό για όλα αυτά που μας είπε. Βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία με την στρατηγική που λέει Trade for All, εμπόριο για όλους. Και εσείς ε, και η προηγούμενη Προεδρία, αλλά και η επόμενη μάλλον θα έχετε αντιμετωπίσει αυτό το πολύ περίπλοκο θέμα. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ορισμένα και βασικά θέματα, τα οποία κατά την άποψή μου έχουν μεγάλη σημασία. Συμφωνώ προφανώς με τους προαλήσαντες για τα ερωτήματα που έθεσαν για τη Συμφωνία ΣΕΤΑ. Αλλά θα ήθελα να μας ενημερώσετε με μεγαλύτερη ακρίβεια το Συμβούλιο Πώς ακριβώς αξιολογεί ε, το σύστημα ISTS, την ε, μετεξέλιξή του. Υπάρχει η ομόφωνη συμφωνία του Συμβουλίου και τι σημαίνει η συμφωνία του Συμβουλίου ε, σε σχέση με την συμπερίληψη αυτής της διαδικασίας σε όλες τις εμπορικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται με τρίτες χώρες. Αυτό πραγματικά με ενδιαφέρει πολύ. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο που με ενδιαφέρει είναι γενικά το Συμβούλιο πώς ακριβώς αξιολογεί τη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Δηλαδή, είναι το Κοινοβούλιο καθοριστικός εταίρος για το Συμβούλιο σε νομοθετικές δραστηριότητες και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο ε, το ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε τον εξυγχρονισμό των ε, διαπραγματεύσεων. Αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τα ε, κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή θεωρούν ότι είναι ε, απόλυτη προϋπόθεση να υπάρξει εξυγχρονισμός του ίδιου του δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εδώ με ενδιαφέρει δική σας η θέση. Όσον αφορά τώρα το πλεονάζον δυναμικών, αυτό το αναφέρεται σε σχέση με την Κίνα. Κοιτάξτε, έχουμε και κάθε ένας από εμά πλεονάζουσες δυνατότητες. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό το Συμβούλιο έτσι ώστε να ε, δρομολογηθεί συνεργασία με την Κίνα και να είναι αποτελεσματική και όχι στο τέλος του έτους να βρεθούμε μπροστά σε ερήπια και να ξεκινήσει εμπορικός ε, πόλεμος. Εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν βλέπω να υπάρχει ελπίδα ακόμα και μετά την τελευταία συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Ε, είπατε ότι το Συμβούλιο ε, θα τοποθετηθεί τον Νοέμβρη για την ε, περίπτωση της ε, ένταξης του Ισημερινού. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ αργά, γιατί στο τέλος του έτους κλείνει η όλη υπόθεση και τότε το Κοινοβούλιο ε, θα είναι αναγκασμένο ταχύτατα να ορίσει τη θέση του. Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι απαραίτητα συμμετοχή των δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων στην εμπορική πολιτική. Πολύ ωραία. Επόμενος ομιλητής. Εκ μέρους των Πρασίνων. Ο κύριος Ζαντό, ευχαριστώ πολύ. Ανακοινώσατε κάποια πράγματα για το, τη συμφωνία ΣΕΤΑ, ότι το θέμα των επενδυτών είναι επίμαχο ε, πώς απειλούνται οι διαφορές δηλαδή κρατών επενδυτών. Ότι δεν θα περιληφθεί στο προσωρινό εφόσον στηρίξει τελικά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αυτή την πρόταση. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω από πλευρά του Συμβουλίου υπάρχει ομοφωνία. Είναι τώρα θέση του Συμβουλίου, έτσι. Η ιδέα ότι η διατησία και οι επενδυτές θα είναι εθνική αρμοδιότητα ή όχι. Ξέρω ότι δεν είναι αυτό η θέση της Κομισιόν. Και νομικά πόσο ισχυρό θα είναι αυτό τη στιγμή που κανονικά το ΣΕΤΑ είναι 100% ε, συμφωνία διεθνής ενώ εμείς θέλουμε να βάλουμε και ένα πολιτικό σκέλος. Πώ θα μπούμε στη διαδικασία επικύρωσης της συμφωνίας αυτής ΣΕΤΑ χωρίς να ξέρουμε τι θα αποφασίσει το δικαστήριο για τη Σιγκαπούρη. Υπάρχει δηλαδή εδώ ένα κενό, μια σάφια. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, είναι μια μεικτή συμφωνία, ναι. Εγώ που είμαι πεπισμένος Ευρωπαίος, δεν μου αρέσει να επαναθνικοποιούμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Οπότε, αν δεν υπάρχει διαφάνεια, η συζήτηση για την παγκοσμιοποίηση στις χώρες μας είναι τέτοια και στα εθνικά κοινοβούλια που πρέπει να συνεχιστεί. Το να λέμε στα εθνικά κοινοβούλια θα συμμετάσχετε στην κύρωση και συγχρόνω να του λέμε ότι έτσι καλώ θα εφαρμοστεί η συμφωνία βάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ένα βαθμό και το Συμβούλιο, χωρί καν εσεί να έχετε προλάβει να κυρώσετε, είναι μια διαδικασία που μα εκπλήσει. Γιατί λέτε, θα έχετε μια αρμοδιότητα, αλλά βάσει τη διαδικασία η αρμοδιότητά σα αυτή κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Εξαιτία της ε, προσωρινή αυτής διευθέτησης. Τέλος, για τον Brexit. Το καλό νέο είναι ότι δεν είναι ο κύριος Μπιν ο οποίος αναλαμβάνει τελικά την Βρετανική διπλωματία. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει να ενεργοποιηθεί το άρθρο 50. Τι θα κάνετε εσείς με το ΣΕΤΑ, με τις ποσοστώσεις κρέατος. Πώς θα διαχειριστούμε τις ποσοστώσεις αυτές από τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο θα έχει ενεργοποιήσει το άρθρο 50 και η εμπορική μας προστασία πώς θα προχωρήσει. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αγωνιστεί πολύ για να μην αφισβητηθούν κάποιες αρχές ότι αποφασίζει αυτός που δικεί. Πώς θα υποστηρίξουμε καλύτερα την Ευρώπη λοιπόν στα πλαίσια αυτά. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Άλλοι τρει έχουν ζητήσει το λόγο. Κρουσβάλτ. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, τα περισσότερα ερωτήματα έχουν ήδη τεθεί. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ που ήρθατε και μας ε, ενημερώσατε και μάλιστα ε, διεξοδικά. Όσον αφορά τώρα στο θεματελόγιο για την εμπορική πολιτική, είναι γεμάτο, πολύ φουσκωμένο. Ε, και εσείς, στην καλύτερη των περιπτώσεων, έχετε μπροστά σας ε, τέσσερις ε, μήνες, εδώ μεταξύ μπαίνουν και πολλές γιορτές. Ξέρετε κάτι, σας εύχομαι καλή επιτυχία και να κάνετε τη δουλειά σας και με ενθουσιασμό και χαρά. Όμως θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η θέση δική σας και του Συμβουλίου. Ανεξάρτητα από όλα αυτά που είπατε για τη Συμφωνία ΣΕΤΑ, μας λέτε ότι ε, δεν θέλετε τη Συμφωνία TTIP, ούτε και εμείς τη θέλουμε. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχουν οι μικτές συμφωνίες, ή μερικές επικυρώσεις, μερικές ε, εφαρμογές. Κοιτάξτε, de facto φτάνουμε σε μία ε, συμφωνία, ομπρέλα, που εμφαρμόζεται σε επιμέρους τμήματα. Ίσως ε, μπορείτε λιγάκι να μας εξηγήσετε πώς ε, τα βλέπετε όλα αυτά και τι προτείνετε να κάνετε συγκεκριμένα κατά τις επόμενες έξι εβδομάδες. Επόμενη μιλήτρια Καρολίνα Κασφάλτερ Χάιντς, παρακαλώ. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Ε, ξέρετε, με ανησυχεί λιγάκι ακούγοντας ε, το θέμα της αγοράς και της Κίνας και ακούω ότι το Συμβουλίο δεν έχει ακόμα καταλήξει, θα περιμένω να δει τι θα αποφασίσει η Κομισιόν. Αλλά ξέρετε, σιγά σιγά πρέπει να αποφασίσει, γιατί το Νοέμβρη εκπνέει αυτή η συμφωνία ΠΟΕ και θα ήθελα να μας πείτε τι πιστεύετε εσείς από αυτής. Γιατί δεν υπάρχει πια αρκετός καιρός και γνωρίζουμε ότι διακυβεύονται πάρα πολλά αν θέλει η Κίνα να διατηρήσει αυτή τη θέση στην αγορά. Πρόκειται για θέσεις απασχόληση, πρόκειται για σημαντικές συνέπειες στο εξωτερικό μας εμπόριο και στην οικονομία μας και θα ήθελα να έχω μια πιο συγκεκριμένη απάντηση εκ μέρου σας για το ποια ακριβώς θα είναι η θέση σας σε αυτό το θέμα. Και τέλος, ο κύριος Μικρομεσαία Επιχείρηση, ο κύριος Ρούμπιχ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως και το εμπόριο παίζει σημαντικό ρόλο ε, για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εμείς επιθυμούμε η παγκοσμιοποίηση να γίνεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Θέλουμε νομική ασφάλεια για τις ΜΜΕ. Άρα δηλαδή οι διαπραγματεύσεις ε, του ΠΟΕ ή τη ΣΕΤΑ είναι ιδιαίτερη σημασία να λαμβάνουν ιδιαίτερη υπόψη οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και στη ΣΕΤΑ και στο TTIP ε, υπάρχει εντολή προς τις 28 κυβερνήσεις και εγώ ερωτώ, οι κυβερνήσεις πώς ακριβώς απέκτησαν αυτήν την εντολή προς διαπραγμάτευση, απευθύνθηκαν στα εθνικά τους κοινοβούλια. Ε, τα εθνικά κοινοβούλια συμμετείχαν κατά την ανάθεση της εντολής και γνωρίζουμε ότι ε, η συμφωνία για τη ΣΕΤΑ έχει ε, εκπληρωθεί μόνο εν μέρη. Δηλαδή δεν έχει ληφθεί υπόψη η στάση των κρατών μελών. Υπάρχει μία ε, συμφωνία επί της οποίας διαπραγματεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα της ε, διευθέτησης διαφορών. Αυτό το διαπραγματεύτηκε εκ των υστέρων ο κύριος Γιούγκερ και έχει κλείσει τώρα και αυτό το θέμα. Και τίθεται το ερώτημα. Οι κυβερνήσεις, τα εθνικά κοινοβούλια θα στηρίξουν αυτά τα οποία έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αν πρόκειται για μεικτή συμφωνία, μήπως εσείς ε, μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς εμπίπτει σε εθνικό επίπεδο, τι πρέπει να ψηφιστεί εκεί και τι είναι εκείνο το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Τώρα που έμπαινα στο Κοινοβούλιο είδα ότι εδώ υπάρχουν ανεβέστατοι λομπίστες κατά του TTIP και το κάνουν αυτό τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν τελειώσει οι διαπραγματεύσεις. Είναι όλα ακόμα ανοιχτά. Και για τη ΣΕΤΑ, ε, ξέρετε, ε, νομίζω ότι στο μέλλον ε, αυτό που θα υπερισχύσει θα είναι φτώχεια για όλους. Εγώ φτώχεια για όλους δεν μ' αρέσει και δεν το θέλω. Ο κύριος Υπουργός. Έχετε την ευκαιρία να απαντήσετε. Τι Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα απαντήσω στα σλοβακικά. Ελπίζω να ακούσετε τη μετάφραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίε και κύριοι, για τις ερωτήσεις σας. Αναφερθήκατε σε αυτά που είπα στην παρουσίασή μου. ΣΕΤΑ, η συμφωνία με τον Καναδά, τη ΤΥΠ, παραχώρηση του καθεστώτος οικονομίας αγοράς στην Κίνα. Αναφερθήκατε στην διαφάνεια, στην συμφωνία με τη Μερκοσούρ. Θα προσπαθήσω σιγά σιγά λοιπόν να καλύψω όλες αυτές τις ερωτήσεις. Σε κάποιους δυστυχώς δεν θα μπορέσω να απαντήσω. Δεν τα γνωρίζω όλα, δεν έχω απαντήσεις για όλα. Ίσως να μην σα ικανοποιήσουν και οι απαντήσει που θα σα δώσω, αλλά τόσο θα προσπαθήσω όσο μπορώ. Για τη ΣΕΤΑ, τη συμφωνία με τον Καναδά. Επαναλαμβάνω ότι η συμφωνία ΣΕΤΑ είναι για μας μια προτεραιότητα στα πλαίσια της γενικότερης εμπορικής πολιτικής της Ένωσης. Επειδή είναι ένας πολύ σημαντικός εταίρος στα πλαίσια του G7. Ο κύριος Ρούμπικ το είπε και αυτός στο τέλος της ομιλίας του, ότι αυτή η συμφωνία συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να υπογράψουμε αυτή τη συμφωνία. Η Κομισιόν την περασμένη εβδομάδα υπέβαλε στο Συμβούλιο μία πρόταση απόφασης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή και την ολοκλήρωση της συμφωνίας ξεκίνησε αμέσω τη δουλειά σε επίπεδο Συμβουλίου η Σλοβακική Προεδρία βάσει αυτών των προτάσεων ώστε να υπογράψουμε την τελική συμφωνία με τον Καναδά τον Οκτώβρη. Εμείς αυτή τη στιγμή δουλεύουμε πάνω στην προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας που είναι απαραίτητη σε σχέση με την αξιοπιστία μας ενώπιον του εταίρου μας του Καναδά. Είναι δύσκολο κανείς να, προβλέψει τα αποτελέσματα αυτής της προσωρινής διαπραγμάτευσης. Δηλαδή τι εύρος θα έχουν οι αποφάσεις, τι θα εφαρμοστεί προσωρινά και τι όχι. Πάντως η προστασία των επενδύσεων και η δικαστική δεν θα είναι αντικείμενο αυτών των προσωρινών αποφάσεων. Αυτό ζητάει η πλειοψηφία των και έτσι θα προχωρήσουν οι συζητήσεις στο Συμβούλιο. Για το TTIP τώρα. Διάφοροι βουλευτές έθεσαν ερωτήματα. Η κυρία Σάκε, πρώτη. Νομίζω ότι και στις δύο όχθες του Ατλαντικού υπάρχει βούληση για την επίτευξη μιας ισορροπημένης και φιλόδοξης συμφωνίας εντός του έτους. Καταφέραμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο σε κάποια θέματα. Παραμένουν όμως κάποια ζητήματα τα οποία δεν έχουν ρυθμιστεί. Πάντως, ο 14ος γύρος διαπραγματεύσεων θα δώσει καρπούς πολύ βασικούς, πολύ σημαντικούς για την τελική ευόδοση της συμφωνίας. Όπως λέγα προηγουμένως, δεν θέλουμε μια συμφωνία light. Θέλω συμφωνία να καλύπτει όλα τα πεδία. Ε, δεν χρειαζόμαστε συμφωνίε δηλαδή απλά και μόνο για να σφίξουμε τα χέρια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλουμε τέτοιε συμφωνίε. Αλλά για αυτά τα θέματα οπωσδήποτε θα συζητήσουμε στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής των Υπουργών Εμπορίου στις 22 και 23 Σεπτέμβρη στην Πρατισλάβα. και όπως και για την συμφωνία ΣΕΤΑ, η TTIP θα συζητηθεί κατά προτεραιότητα, όπως επίσης κατά προτεραιότητα θα συζητηθεί και το θέμα της απόδοσης της οικονομίας αγοράς στην Κίνα. Υπήρξαν διάφορες ερωτήσεις επί τη ευκαιρία σχετικά με την Κίνα. Το έθεσε το θέμα ο κ. Βίνκλερ, Ζαχραντήλ, επίσης και ο κ. Χάιντς. και εσείς μιλήσατε για αυτό το θέμα της Κίνας. Νομίζω πάντως ότι το γεγονός είναι ότι δεν έχουμε ακόμα μια οριστική πρόταση της Κομισιόν. Δηλαδή το Συμβούλιο και αυτό δεν έχει ακόμα οριστική θέση σε σχέση με την απόδοση του καθεστώτος οικονομίας αγορά στην Κίνα. Κύριε Χάιντς, με ρωτήσατε πώς γίνεται αυτό. Τι να σας πω εγώ, εδώ και μια εβδομάδα έχω αναλάβει ε, τώρα τι γίνεται στο Συμβούλιο ή τι γινόταν πριν, δεν ξέρω τι να σας πω. Πριν από εμά είχαμε τους Ολλανδούς. Ε, υπό τους Ολλανδούς δεν είχαμε μια τελική πρόταση, μια πρόταση συμφωνίας. πάντως στόχος μας είναι να υποβάλει μια πρόταση κομισιόν στο Συμβούλιο, κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί και από τη στιγμή που δεν έχει συμβεί, δεν έχουμε κάποια βάση πάνω στην οποία θα κάνουμε αξιολόγηση και θα υποβάλουμε τη δική μας πρόταση. Πάντως, για αυτό το θέμα της απόδοσης του καθεστώτος οικονομίας αγορά στην Κίνα νομίζω ότι ίσως η τελική απόφαση να μην προέλθει από τους Υπουργούς Εμπορίου ίσως να προέλθει από υψηλότερο επίπεδο καταλαβαίνετε γιατί στα θέματα εμπορίου εμπίπτουν και πολιτικά ζητήματα οπότε ίσως χρειαστεί απόφαση από υψηλότερο επίπεδο κάποιος ε, με ρώτησε πώς όλη αυτή η διαδικασία επηρεάζει την ίδια τη Σλοβακία και τα μέτρα προστασίας. Εμείς οπωσδήποτε θα έχουμε επιπτώσεις από αυτή τη συμφωνία με την Κίνα. Έχουμε ισχυρή χαλιβουργία και οι τιμές οι οποίες είναι αντικείμενο, μάλλον αποτέλεσμα του dumping, πραγματικά αποτελούν μια απειλή για μας, για τη μηχανία της χώρας μας. Πάντως, εμείς έχουμε ξεκάθαρες ιδέες τι θέλουμε να κάνουμε, όμως θα προσπαθήσουμε να τα διαχωρίσουμε αυτά από την πορεία της Προεδρίας μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτό το εξάμεινο και θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο πιο ισορροπημένοι γίνεται και ακριβοδίκαιοι για αυτά τα θέματα. Τώρα, για την εντολή των διαπραγματεύσεων. Είχαμε διάφορες ερωτήσεις εδώ για αυτό το θέμα. Σχετικά με τις δεσμεύσεις όσον αφορά την τακτική και διαφανή ενημέρωση του Κοινοβουλίου κατά διάρκεια όλων αυτών των διαπραγματεύσεων και σε σχέση επίσης με τις εμπιστευτικές πληροφορίες, το Συμβούλιο θα αξιολογήσει τα θέματα αυτά αναπερίπτωση. Δηλαδή αναπερίπτωση θα αξιολογήσει τα αιτήματα του Κοινοβουλίου για εμπιστευτικές πληροφορίες, υπαρχή εμπιστευτικών πληροφοριών και κοινοποίηση του περιεχομένου των εντολών για τις διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία με το Μεξικό ήδη έχουμε διαβιβάσει το αίτημα για πληροφορίες στην Κομισιόν και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται βέβαια για να στέλνουμε πληροφορίε σχετικά με την εντολή διαπραγμάτευση που αφορά το Μεξικό. Χθες το Κορεπέρ έδωσε το πράσινο φως για την άξιση των διαπραγματεύσεων με την Ινδονησία. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν στο Συμβούλιο να βρούμε μια συμφωνία γρήγορη ώστε να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει και για την περίπτωση της Τινησίας, για το ελεύθερο εμπόριο με την την Ισία. Το ίδιο έκανε παλαιότερα και το Συμβούλιο για άλλες διαπραγματεύσεις, TTIP και άλλες συμφωνίες. ΣΕΤΑ Πάντως πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι οι διαπραγματεύσεις των εμπορικών συμφωνιών απαιτούν κάποιο, κάποια εμπιστευτικότητα ακριβώς για να διασφαλίσουμε το περιεχόμενο αυτών των διαπραγματεύσεων. Καταλαβαίνω βέβαια ότι εσείς έχετε κάποιες ανησυχίες ή αφιβολίες. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν εσείς έχετε εργαστεί στον εμπορικό τομέα κατά διάρκεια της επαγγελματικής σας ζωής, αλλά τέλος πάντων όταν κάποιος κάνει διαπραγματεύσει ας για να αγοράσει ένα οικόπεδο, ε, δεν θα πάει να κοινοποιήσει τέλος πάντων το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης για την αγορά πολισία. Αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και με αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι συμπαγής σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ε, θα πρέπει να ενεργεί με μια φωνή, ώστε να πετύχει και τα απαραίτητα εμπορικά πλεονεκτήματα. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι η κοινοποίηση, η δημοσίευση εμπιστευτικών εγγράφων σημαίνει ότι παρακάμπτουμε το Κοινοβούλιο. Είναι ένα θέμα στρατηγικής απλά και μόνο στα πλαίσια της διαπραγματεύση Πάντως, Πάντως θα έχετε πρόσβαση στα έγγραφα όταν αυτά βέβαια τα έγγραφα δεν θα έχουν επιπτώσεις στην στρατηγική των ίδιων των διαπραγματεύσεων. Τώρα για τη χιλή. Είχαμε μια ερώτηση σχετικά με αυτή. Η Σλοβακία είναι υπέρ του εξυγχρονισμού της συμφωνίας με τη Χιλή που ανάγεται στο 2003. Κάνει και μια αξιολόγηση αντικτύπου εσωτερική η Κομισιόν και νομίζω ότι στη συνέχεια θα μπορούσε να υποβάλει μια πρόταση εντολής για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει το 2017. Κατά τη διάρκεια της Σλοβακικής Προεδρίας δεν προβλέπουμε ακόμα την εντολή, την ολοκλήρωση της εντολής για την Χιλή. Πρόεδρε, προσπάθησα να απαντήσω στο, στην πλειοψηφία τουλάχιστον των ερωτήσεων που μου θέσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Once again, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα να συζητήσουμε μαζί τις προτεραιότητες της Προεδρίας σας. Είπαν και οι συνάδελφοι, εδώ είναι πολύ φιλόδοξο το πρόγραμμά σας. Σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο λοιπόν. Καλή τύχη σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Υπάρχει και το Brexit και πολλά άλλα δύσκολα σημεία που έχετε στην ημερήσια διάταξή σας. Ευχαριστούμε λοιπόν και θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε. Dear, Αγαπητοί συνάδελφοι, πάμε λοιπόν τώρα στις ψηφοφορίε και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω ότι οι ψηφοφορίες γίνονται ονομαστικά ε, και γι' αυτό χρειαζόμαστε την κάρτα. Θα ήθελα λοιπόν ε, να σας παρακαλέσω να βγάλετε την κάρτα σας, να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Και ε, κάνουμε τώρα τη δοκιμαστική ψηφοφορία. Liebe Kollegen, stimmen Sie bitte ab. Ψηφίζουμε λοιπόν.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 Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω μαζί μου την κάρτα, την ξέχασα, θα μου τη φέρουνε, γι' αυτό θα ψηφίζω ψώνοντα το χέρι. Λυπάμαι, τι να κάνω. Εντάξει, δεν πειράζει. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν στην πρώτη ψηφοφορία. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της τριμερούς συζήτησης για τα torture goods μπορεί ορισμένων δικημένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή απάνθρωπη κτλ. Ψηφίσαμε στις 23 Μαΐου και τώρα έχουμε το τελικό κείμενο αφού εξετάστηκε ε, βελτιώθηκε γλωσσικά, νομικά. Φαντάζομαι ότι το έχετε δει και θα έχετε διαπιστώσει ότι ως Κοινοβούλιο ε, σημειώσαμε μεγάλη επιτυχία όσον αφορά αυτή την ε, νομοθετική ρύθμιση. Και γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε την εισηγήτριά μας, την ε, Μαρίτε Σάκε, που ε, ήταν επικεφαλής των διαπραγματεύσεων. Μαρίτε, θέλεις να πεις κάτι? Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω πολλά. Ευχαριστώ απλώ τους συναδέλφους για τη συνεργασία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Αρχίζουμε λοιπόν με την ψηφοφορία τότε. Μία ψηφοφορία έχουμε για αυτό το θέμα, ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα της ψηφοφορίας. Ωραία, εγκρίθηκε. Τώρα, το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε αυτό το θέμα. Και θα έπρεπε να ζητήσουμε συζήτηση στην Ολομέλεια για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε και στο κοινό τις απόψεις μας. Καλώς. Ωραία. να ρωτήσω τι ψηφίσατε, υπέρ ή κατά. Αποχή. Could I make a point of order, please? Ε, έχω διαδικαστικό. Μπορεί κανείς να βρει μια κάρτα στο κτίριο. και στις Βρυξέλλε και στο Στρασβούργο μπορείτε να ζητήσετε κάρτα για να ψηφίσετε. Γίνεται. Κυρία Μπιτζότο. Ευχαριστώ. Das äh, mit äh, Εδώ λοιπόν είναι η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ε, με τις χώρες ΟΕΣ και τις ΚΑΜΑ κτλ. Ε, συγητής ο κύριος Λάμστοφ ε, και υπάρχει μία σειρά τροπολογιών που δεν έγιναν αποδεκτές, όμως μπορούμε να ψηφίσουμε για την υπαρχμόν δύο. Και ποιο συμφωνεί παρακαλώ με την δύο. κατά, υπερκατά, αποχές, απορρίπτεται. Και πάμε την ηλεκτρονική τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Η Abstimmung ist geschlossen. 22. Έκλεισε η ψηφοφορία 22 υπέρ και ε, 9 κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια κύριε Λάμπστορ. Dann kommen wir zu einem wundervollen Bericht. Πάμε τώρα σε μια θαυμάσια έκθεση για τις εξωτερικές εμπορικές ε, ε, στατιστικές. Είναι μια ιστορία που ελπίζω να κλείσει σήμερα, γιατί το Συμβούλιο σε αυτό το θέμα δεν επέδειξε ευελιξία. Αλλά τώρα έχουμε ένα κοινό κείμενο το οποίο αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα της ε, τριμερούς ε, συζήτησης. Και ξεκινάει η ψηφοφορία σχετικά με αυτές τις εξωτερικές στατιστικές. Λοιπόν, Ψηφίσαμε, ψηφίσατε φαντάζομαι. Έχετε όλη κάρτα ψηφοφορίας, 30 υπέρ και τρεις αποχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 18. Πρόκειται για τη διεύρυνση της συμφωνίας με την Κίνα, ε, να περιληφθεί και η Κροατία. Ξεκινάει λοιπόν η ψηφοφορία. Έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίθηκε και αυτό με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κυρία, κύριε Μπίνκλα. Και πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 19 Πρόκειται για την προσθήκη της συμφωνίας ΓΚΑΤ ε, να προσθεθεί και η Κροατία. Και εδώ λοιπόν ψηφίζουμε Έκλεισε η ψηφοφορία. Πάλι 31 υπέρ. Και πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 20. Πρόκειται για το μέλλον. Μάλλον ξέχασα να σε χαρώ τον κύριο Τσάλμπα. Συγχαρητήρια. Πάμε στο 20. Το μέλλον των σχέσεων ε, ΑΚΕ, χωρών ΑΚΕ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά το 2020, μετά την ε, εκπνοή της Συμφωνίας Κοτονού. Πάμε. Τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την υπαριθμόν 1. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2. Ένα, λέει ο πρόεδρος, συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 8. Προσθήκη της 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Πάμε στην τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ για την 14. Ε, ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλεισε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Η 15 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα ηλεκτρονική επαλήθευση για τη 15. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 16. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 22, πρώτο τμήμα παρακαλώ, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η τροπολογία 26 για το δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 30 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η 31 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ. Ε, ε ελέγχουμε για την 31 ψηφίζουμε παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στη 40. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 41. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 42. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται η 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Η 4α συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 57 παρακαλώ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 59 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 66 υπέρ κατά αποχές Μισό λεπτό, ηλεκτρονική επαλήθευση για την 66. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Και έκλεισε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Η 67 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και Περνάμε στο, στην τελική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Και κλείσει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια Πέντρο. Πάμε τώρα στο υπαριθμόν 21 σημείο είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έναντι του Ιράν σε συνέχεια της πυρηνικής συμφωνίας και έχουμε καταρχήν τη συμβαστική πρόταση 1 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται θα μπορούσε να ε, υπάρχει προσθήκη στη, με την τροπολογία υπερθμών 1 υπέρ κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να έχουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία υπαριθμών 1. Ψηφίζουμε, παρακαλώ. Έκλειση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Η συμβαστική 17, υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση παρακαλώ, για την 17. Ψηφίζουμε. Έκλειση ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 18. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 25 ως ε, ενδεχόμενη προσθήκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίζουμε παρακαλώ έκλεισε ψηφοφορία πράγματι απορρίφθηκε Συμβιβαστική 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 32 Συγγνώμη, σκέτη τροπολογία δηλαδή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 39 καταπίπτει. Και κατόπιν τούτου πάμε στην 45. Υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την 45 υπέρ. Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά. <laughs> Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, μπερδεύτηκα, λέει ο Πρόεδρος. Έκλεισε η ηλεκτρονική ψηφοφορία και όπως σας είπα εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 51 υπέρ, κατά, Συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος, λάθος έκανα. Για την 52 ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η τροπολογία 55 η 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 57 σε δύο τμήματα ψηφίζουμε. Για το πρώτο τμήμα παρακαλώ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Για το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε, τελική ψηφοφορία, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε παρακαλώ. Abstimmung Έκλεισε η ψηφορία και εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια. Θερμά συγχαρητήρια. Και πάμε τώρα στην τελευταία ψηφοφορία για σήμερα είναι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και παρακολούθηση από την κοινωνία των πολιτών της ε, Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΜΑ. Εδώ υπάρχει μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ψηφίζουμε παρακαλώ. Und die Abstimmung ist geschlossen und ist auch hier mit großer Και αυτό εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Κατόπιν τούτου ψηφίσαμε, πάει, τελειώσαμε ε, με τις ψηφοφορίες, τα ξεπετάξαμε σε μισή ώρα. έτσι. Αγαπητοί συνάδελφοι, Κάποιοι συνάδελφοι, παρόλο που για μένα δεν έφτασαν ακόμα καλοκαιρινέ καλοκαιρινές διακοπές, κάποιοι φαίνεται ότι θέλουν να αποχωρήσουν. Ισύχω, παρακαλώ. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το σημείο για την παρακολούθηση δραστηριοτήτων ομάδων. Αυτή η άσκηση, η παρακολούθηση δηλαδή δραστηριοτήτων ομάδων είναι ένα ενδιαφέρον θέμα. Τους τελευταίους μήνες είχαμε δραστηριοποιηθεί πολύ για την παρακολούθηση αυτή. Είχαμε 17 συναντήσεις παρακολούθησης δραστηριοτήτων ομάδων, κάτι το οποίο δείχνει ότι είμαστε πραγματικά δραστήριοι. Τώρα τι θα μπορούσε να βοηθήσει, είχαμε για τις ΗΠΑ, για την TTIP, τέσσερις συναντήσεις, 19 Απριλίου συγκεκριμένα, με τον ε, δεύτερο στις διαπραγματεύσεις και τον 13ο ε, γύρο και μετά στις 3 Μαΐου τον Ιγνάσιο 29 Ιουνίου είχαμε την, ε, το σχέδιο μελέτης για τις προδιαγραφές και τις ρυθμίσεις αξιολόγηση κινδύνου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά ήταν πολύ ενδιαφέροντα και βέβαια προετοιμαστήκαμε και στις 13 Ιουνίου για τον 14ο γύρο. Μετά το καλοκαίρι αμέσως θα έχουμε και πάλι συνάντηση για την προετοιμασία του 14ου γύρου. Συνεπώς, κλείνουμε για τις διαπραγματεύσεις και είναι σαφές ότι θα συζητήσουμε την αξιολόγηση για το 14ο γύρο μετά το καλοκαίρι. Κεντρική Αμερική και Κούβα τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είχαμε μία συνάντηση, λέει ο κύριος Μπάγκια, με την πρεσβεία της ε, Κούβας, την παρουσία της Γενικής Διεύθυνσης Trade. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει, χωρίς να μας πει γιατί. Και θα ήταν ενδιαφέρον να ήταν εκεί, γιατί η συζήτησή μας επικεντρώθηκε στον πολιτικό διάλογο και τη συμφωνία συνεργασίας. Η πρέσβης πρώτον ζήτησε να σταματήσει πια ισχύει η κοινή θέση του 1996 και επέμεινε ότι η διαδικασία του εμπόριου, ο διάλογος για το εμπόριο, η ένταξη της Κούβας στην παγκόσμια οικονομία είναι ο στόχος, αλλά όχι συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ούτε για τώρα ούτε για το μέλλον. Αυτό ήταν ένα σαφές μήνυμα. Η Γενική Διεύθυνση Trade είπε ποια είναι η κατάσταση μέχρι τώρα στο διάλογο αυτό και τη Συμφωνία Συνεργασίας. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι η Κούβα δεν μπορεί να επωφεληθεί πια από τη Συμφωνία GSP. Υπάρχουν βέβαια πολύ ενδιαφέρουσε εξελίσει στην Κούβα, στην οικονομία της δηλαδή. Για παράδειγμα, αυτοαπασχολούμενοι. Επίσης, 5% των τροφίμων που παράγει η χώρα βασίζεται στο 28% του εδάφους της, της επικράτειας. Είναι ενδιαφέρον αυτό να το λάβουμε υπόψη μας για την εξέλιξη της οικονομίας. Όσον αφορά το PDCA, προς το παρόν έχουμε 18 διμερείς επενδυτικές συμφωνίες, Κούβα, Ενωμένες Πολιτείε. Υπάρχει μια νέα συμφωνία που ολοκληρώθηκε, που δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα. Τα συμπεράσματα θα τα έχουμε τέλος του 2016, αρχές του 2017. Και έπειτα όλοι γνωρίζουμε και την ε, συνήθη κατάσταση που επικρατεί στη διαδικασία επικύρωσης. Βέβαια, η Κούβα σίγουρα θα προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα από την Ευρώπη και εδώ. Είναι όμως μια πρόκληση. Να μην μιλάμε μόνο για την Συμφωνία ΣΕΤΑ, το TTIP. Είχαμε συνάντηση και με πρέσβεις από τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής που επέμειναν και μας πίεσαν σε επίπεδο συμβουλίου να πούμε ότι οι χώρες μέλη πρέπει να κυρώσουν πιο γρήγορα τα βάζουν με εμά. Θέλουμε πάνω από δύο χρόνια για να κυρώσουμε τέτοιε συμφωνίε ενώ υπάρχει ομοφωνία όσον αφορά το περιεχόμενο. Δεν δικαιολογείται, δεν εξηγείται. Θα υπάρχουν και κεφάλαια για τον πολιτικό διάλογο, τη συνεργασία και την εμπορική συνεργασία. Δεν είναι συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, όπως είπαμε. Παραμένουν ζητήματα, κάποιοι στόχοι του ΠΟΕ δύο συνεργασία σε τασμολογικά εμπόρια, τελωνία κλπ. Και υπάρχει και ένα ειδικό άρθρο για τις επενδύσεις, για να υπάρχει ένα προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον. Αυτά περιλαμβάνει η συμφωνή και φυσικά και μια ρήτρα αναθεώρησης. Ήταν ένα ενδιαφέρον σημείο κίνησης. Ο δρόμος θα είναι μακρύς όμως. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Όντως, it's a long way to tip away, λέει ο πρόεδρος. Σαντακ. 26 Απριλίου είχαμε τη συνάντησή μας. Η Σαντακ είπα, συζητήθηκε και εγκρίναμε συμφωνία. Η Ιαπωνία, 3 Μαΐου. Όπως είπε και ο εκπρόσωπος της Σλοβακικής Προεδρίας Υπουργός, εκεί τα πράγματα πάνε αργά γιατί υπάρχουν εκλογές στην Ανοβουλή εκεί. Και την προηγούμενη εβδομάδα ή την προπροηγούμενη προχωρήσαμε. Ελπίζουμε τώρα να μπορέσουμε να επιταχύνουμε μετά από τις εκλογές αυτές. 27 Ιουνίου είχαμε άλλη συνάντηση μετά το διαπραγματευτικό γύρο 14 και κάποιοι παράγοντες συμμετέχουν, όπως για παράδειγμα ο κλάδος κατασκευής ποδηλάτων, ποδηλατοδρομίας. Και όπως είπα και χτες, είμαστε σε καλό δρόμο. Μαγκρέμπα, 24 Μαΐου. Πολύ υποσχόμενο ο πρώτος γύρος και των διαπραγματεύσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ισίας. Είμαι πεπισμένο ότι είναι ένα σημαντικός φάκελος αυτός και ότι μπορούμε να στηρίξουμε τις εξελίξεις στην Τινησία. Τίζα. Δύο ομάδες παρακολούθησης είχαμε, 21 Μαΐου και 30 Ιουνίου. Μετά το 17ο και 18ο γύρο διαπραγματεύσεων. Θα θυμόσαστε την τελευταία φορά, εδώ συζητήσαμε με την κυρία Ρέντινγκ, την εισηγήτρια για τις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τη Συμφωνία Τίζα. Νότια Ασία. 30 Μαΐου είχαμε παρακολούθηση ομάδας. Συζητήσαμε τα εργασιακά δικαιώματα, ε, Διεθνής Γραφείο Εργασίας και διάφορα άλλα. Θέλουμε την εφαρμογή συμφωνίας με τον Μπαγκλαντές. Συζητήσαμε πρωτοβουλία και την περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό. Η Επιτροπή όλο και προετοιμάζεται. Θα μας φέρει ένα καλό αποτέλεσμα φαντάζομαι αφού κρατάει τόσο. Και το GSP-SYN για το Σρι Λάνκα. Και αυτό περιμένουμε. Μολδαβία. 31 Μαΐου είχαμε συνάντηση. Συζητήσαμε στις 29 Ιουνίου το Μερκοσούρ Ή προσφορά για πρόσβαση στην αγορά στο Μερκοσούρ. Μια καρποφόρα προσπάθεια ήταν και αυτή. Μετά, είπα, ομάδες παρακολούθησης για την Ανατολική Αφρική και Δυτική Αφρική. Συμφωνίε εταιρική σχέσης, 12 Ιουλίου. Έλμοντ, μήπως έχεις εσύ να προσθέσεις κάτι σε αυτά. Κοιτάξτε κύριε Πρόεδρε, εχθές είχαμε μία ε, σε βάθος ανταλλαγή απόψεων ε, για την Αφρική, έτσι σε γενικές γραμμές και τα προβλήματα που συζητήσαμε χθες, ε, τα θέματα αυτά ξεκινάνε και από την εξή βάση. Τι θα κάνουμε με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τι θα κάνουμε με τη δυνατότητα να συζητήσουμε για οικονομικές συμφωνίες με τις χώρες της Αφρικής. Ανθρώπινα δικαιώματα και οικονομικές συμφωνίες. Αυτό λοιπόν αυτή η αντίφαση προέκυψε όσον αφορά το θέμα των χωρών της Ανατολικής Αφρικής. Και είχαμε προσκεκλημένους και την Κομισιόν και ΜΚΟ. Ο καθένας ε, είπε βέβαια τη δική του άποψη σχετικά με τη σύναψη συμφωνιών. Είχαμε και εκπροσώπους από την Κένια, την Ουγκάντα και τη Ρουάντα και νομίζω ότι η ανταλλαγή απόψεων ε, της ομάδας monitoring ήταν πολύ σημαντική για να συνεχιστούν εργασίες για τη σύναψη συμφωνίας. Εγώ πιστεύω ότι τελικά πρέπει λιγάκι να παρακολουθήσουμε το κατά πόσο οι χώρες αυτές είναι πρόθυμες να συνάψουν τη συμφωνία. Γιατί ξέρετε κάτι εντυπωσια το γεγονός ότι η Τανζανία δεν φλέγεται και δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Γι' αυτό λοιπόν ας περιμένουμε να δούμε, να δούμε τελικά ε, τι θα γίνει με την ε, σύναψη σχέσεων με τις ε, χώρες της Ανατολικής Αφρικής και πώς μπορούμε τις σχέσεις αυτές να τις τεκμηριώσουμε και με συγκεκριμένη συμφωνία. Πολύ ωραία. Είχαμε λοιπόν την Monitoring Group για Ασία, Φιλιππίνες, Ινδονησία. 12 του μηνός συνεχίζονται διαπραγματεύσεις με τις Φιλιππίνες και σε αυτήν την ομάδα παρακολούθησης συζητήθηκε ο πρώτος γύρος και είναι πολλά υποσχόμενο το χείρημα αυτό με τις Φιλιππίνες. Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίζει και τις ε, διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινδονησίας. Πολλές λοιπόν διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα καταφέρει να έχει δηλαδή στη διάθεσή της τα μέσα να προχωρήσει με τις διαπραγματεύσει αυτές. Και τέλος, ένα από τα καυτά ζητήματα, η καυτή πατάτα, η Κίνα. Συνομιλίες με την Κίνα είχαμε τις τελευταίες μέρες. Το θέμα της απόδοσης του καθεστώτος της αγοράς είναι ένα καυτό και ο Σβίγκλερ είναι ο εισηγητής μας και θα του δώσω και το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είχαμε αυτή τη βδομάδα την ομάδα. Δεν επικεντρωθήκαμε όμως στην απόδοση του καθεστώτος αυτού αγοράς. Αλλά συζητήσαμε για επενδύσεις με την Κίνα. Σε αυτό επικεντρωθήκαμε. Έχουμε ήδη 11 γύρους διαπραγματεύσεων με την Κίνα για επενδυτική συμφωνία, που είναι μια συνολική συμφωνία για επενδύσεις, έτσι ονομάζεται. Comprehensive Agreement for Investments. Ενημερωθήκαμε λοιπόν για το περιεχόμενο της πρότασης από τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κύριο Λέκοβιτς, και θα συζητήσουμε ανταλλαγή προσφορών και πρόκειται για μια μεικτή προσέγγιση. Σε εθνικό επίπεδο θα υπάρχει ένας αρνητικός κατάλογος και για την πρόσβαση στην αγορά θα υπάρχει ένας θετικός κατάλογος. Οι προσφορές αυτές θα συζητηθούν και ελπίζουμε όλοι ότι το Σεπτέμβριο θα τα καταφέρουμε. Για τη διάσκεψη κορυφής με την Κίνα θα αποφασίσουμε τώρα αυτές τις μέρες. Πρόθεσή μας πάντως είναι το Σεπτέμβριο να οργανωθεί ο 12ος γύρος συζητήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει μια μελέτη αντικτύπου που θα είναι ενδιαφέρουσα και για τη δικιά μας Επιτροπή αλλά και για ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα υπάρξει προσωρινή έκθεση για την αξιολόγηση αυτή που θα αναθεωρηθεί και σύντομα. Την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο θα είδατε ότι είχαμε τη νέα στρατηγική για την Κίνα. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ετοίμασαν. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι πάντα τα μηνύματα που παίρνουμε από τον επιχειρηματικό μας κόσμο, τις επιχειρήσεις μας οι εξελίξεις είναι ανησυχητικές στο επιχειρηματικό κλίμα, γιατί οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν μας στέλνουν τα καλύτερα δυνατόν ε, σήματα, μηνύματα. Υπάρχουν και εξωτερικοί παράγωγες, η εισαγωγή άλλων ε, τακτικών για νέες συνθήκες, στην Κίνα για παράδειγμα, κάτι το οποίο δεν είναι καλό σημάδι. Έχουμε και τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων στην ομάδα παρακολούθησης, αλλά και τεχνικούς παράγοντες από πλευρά στην Κίνα, τον κύριο Τσάι, και καρποφόρο διάλογο μαζί τους, παρόλο που πολλά στοιχεία παρέμειναν γενικά όσον αφορά τη θέση της Κίνας. Η, η κυρία Τσάι μας ε, παρουσίασε τις θέσεις της, αλλά πέφυγε να απαντήσει συγκεκριμένες ερωτήσεις μας, γιατί είπε ότι δεν αποτελεί μέρος της διαπραγματευτικής ομάδας των Κινέζων. Πάντως εμείς λέμε τις προτάσεις μας, οι Κινέζοι λένε να μην είναι σε διμερή επενδυτική συμφωνία, αλλά σε FTA, δηλαδή συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Ε, αυτά είναι ευαίσθητα για μας ζητήματα συζητήσαμε και για την Προεδρία του G20 για τις συμφωνίες επίσης διευκόλυνσης και κάποιες φιλοσοφικές ε, ιδέες για την Κίνα, η οποία θέλει να μας πει ότι περιφερειακές συμφωνίες πολυμερείς, όπως TTIP ε, και τα λοιπά, κατά την άποψη των Κινέζων μπορεί να έρχονται σε αντίφαση με τις πολιτικές μας των ΠΟΕ. Έτσι κι πάντα με τους Κινέζους πρέπει να έχουμε και φιλοσοφικές συζητήσεις. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, αφού θα υπάρξει γύρω στην... το Σεπτέμβριο, θα σας ενημερώσουμε μετά. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Δύο διαφορετικές ερωτήσεις. Την πρώτη αναφέρατε για τη Στριλάνκα. Να μας πείτε κάτι παραπάνω. Έστω και δεν έχετε να πείτε τίποτα. Για την Κίνα. Υπάρχει μια ανησυχία μεταξύ των ψηφοφόρων μου ότι αυτό το καθεστώς θα περάσει για την Κίνα και την οικονομία αγοράς σύντομα και θα έχει τεράστιες επιπτώσεις μακροπρόθεσμα αλλά και βραχυπρόθεσμα. Κύριε Βίνκλερ, μπορείτε να σχολιάσετε γι' αυτό. Νομίζω είναι μια ησυχία που μοιράζονται και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, έστω και αν ενδιαφέρονται και τόσο για αυτά που να αποφασιστώ. Ναι, για τη Στριλάνκα. GSP συν. Μέσω κατεξουσιοδότηση πράξης πρέπει να γίνει. Να δούμε τώρα αν αυτές 27 προϋποθέσεις στηρούνται ή όχι. Αυτό συζητιέται. Δεν έχουμε καταλέξει ακόμα για κάποιες πτυχές όπως περιβάλλον, ε, εργασιακά κτλ. Για την Κίνα, ναι, να σας πω ότι και οι δικοί μου ψηφοφόροι μοιράζονται τις ανησυχίες για την απόδοση καθεστώτος οικονομίας αγοράς στην Κίνα. Και είναι σαφές επίσης ότι πριν από λίγο είχαμε ψήφισμα στο Κοινοβούλιο που ήταν σαφέστατο εμείς λέμε στο ψήφισμα ότι θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει κάποια μυντικά εργαλεία για το εμπόριο μετά την 1η Δεκέμβρη. Τα είπα αυτά το Κοινοβούλιο και κυρίως για την χιλιβουργία που είναι πιο ευαίσθητη και άλλες βιομηχανίες όμως. Τώρα, ο λόγος είναι στην Κομισιόν. Το Κοινοβούλιο τοποθετήθηκε, τώρα είναι σειρά της Κομισιόν. Και αν δείτε τι είπε χθε στο Πεκίνο ο Μάστρο, η Μάστρομ και ο Γιουνκέρ, τότε την επόμενη εβδομάδα στις 20 του Ιούλη δεν θα έχουμε ακόμα πρόταση από την Κομισιόν. Είχαν κάποιες διερευνητικές επαφές και δεν θα έχουμε ακόμα την επόμενη εβδομάδα πρόταση. Αλλά το μήνυμα ήταν σαφές τι είδο δηλαδή πρόταση προσδοκούμε από την Κομισιόν για το PDI και τέλος πάντων κάτι το οποίο θα είναι καλό για όλους. Ο Χέλμοντ. Ναι. Να μην ξεκινήσουμε τα συζήτηση. Έχουμε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου και εντάξει το ξέρουμε. Ξέρουμε τι λέει. Αλλά μια και μιλάτε για τους φόρους σας να πείτε τότε στους Βρετανούς ότι η Βρετανική, μια Βρετανική κυβέρνηση επέμενε για τον εξοχρησμό αυτού του εργαλείου άμυνας για δύο χρόνια. Οπότε όλε οι 28 κυβερνήσει θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο. Αυτό πρέπει να υποθεί και να είναι ξεκάθαρο. Αν μιλάμε για διαφάνεια, και σαφήνεια για το ποιος αποφασίζει τι και σε τι επίπεδο, τότε αυτά πρέπει να υποθούν και να καταλάβουν οι πολίτες τι κάνει η Ένωση, τι πολιτικές ακολουθεί. Γι' αυτό ακριβώς θα σας ζητήσω να πείτε στους πολίτες και στους ψηφοφόρους σας συγκεκριμένα πράγματα και να τους ζητήσετε να πιέσουν και τη Βρετανική κυβέρνηση μελλοντικά για αυτή την κατάσταση. Να απαντήσω Άμεση ερώτηση και καλή ερώτηση έτσι. Καταρχάς, μέχρι τώρα η Βρετανική κυβέρνηση δεν έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εγώ δεν είμαι μέλος της κυβέρνησης, ανήκω σε άλλο κόμμα. Αλλά το να κανεί κανείς τα χέρας του δεν είναι και τόσο καλό. Δεν είναι καλή απάντηση. Κάνει τελείως λάθος νομίζω η Βρετανική κυβέρνηση σε αυτό το θέμα και η πολιτική για την Κίνα ήταν το χαρακτηριστικό της πολιτικής, της πορείας πολιτικής του Τζος Όσμπορν, του προηγούμενου Υπουργού Οικονομικών που έφυγε, τον έδιωξαν και ο Λίαν Φόξ, ο Δόκτωρ Λίαν Φόξ θα είναι ο νέος Υπουργός Εμπορίου και θα έχουμε και νέο Υπουργό Οικονομικών και ελπίζω να ακολουθήσουν την άποψη που έχουν όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου ότι οι Κινέζοι κάνουν ντάμπιγκ ιδιαίτερα στην τομέα του χάλιβα. Αν λοιπόν λάβουν το καθεστώς οικονομίας αγοράς οι Κινέζοι, τότε θα είναι πολύ πιο δύσκολο να υιοθετήσουμε τα απαραίτητα αμυντικά μέτρα για το εμπόριο. Οπότε, από τη συνάλφα και σε συντονιστά, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να μεταφέρω τα κέρια σου σχόλια στη Βρετανική κυβέρνηση. Είχαμε όμως βασική σημαντική αλλαγή σε πολιτικό προσωπικό. Ελπίζω να υπάρξει αλλαγή αντίστοιχη σε πολιτικές. Α, βλέπω μια νέα συμμαχία εδώ στο Βούλιο. Νομίζω ότι αυτή τη συζήτηση μπορούμε να την ξαναξεκινήσουμε μετά τις ε, καλοκαιρινές διακοπές, διακοπές στις 20 Ιουλίου. Η Κομισιόν θα, θα συζητήσει για αυτό το θέμα και μετά τις ε, καλοκαιρινές διακοπές, αρχές Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι η Κομισιόν ε, θα καταθέσει μια πρόταση. Helmut. Κοιτάξτε, δεν θέλω να καθυστερήσουμε και να μακρηγορήσω, αλλά θέλω να πω στον συνάδελφό μου, κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ακριβείς. Και εάν υπάρχει πλειοψηφία σε ενδικά χέρια για αυτά τα προγράμματα σε σχέση με το Χάλιβα, ε, θα πρέπει να μας πείτε τι ακριβώς κάνουν ε, για να εξυγχρονίσουν την παραγωγή χάλιβα σε ανώτατο επίπεδο. Είναι και αυτό θέμα dumping. Το θέμα είναι ότι αν δεν βελτιώσει κανείς τις ικανότητές του για να ε, προσαρμοστεί στον εξυγχρονισμό, οι Κινέζοι εξυγχρονίζονται και έχουν περιορίσει και αυτοί την παραγωγή του χάλιβα. Το θέμα είναι πιο περίπλοκο. Δεν φτάνει να πει κανείς ότι ε, οι Κινέζοι κάνουν ε, dumping. Ο ελάχιστο μισθό στην Κίνα είναι υψηλότερο από ό,τι στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Το θέμα είναι ε, το πώς μπορούμε να δούμε τη συνεργασία με τρίτες χώρες και αυτή να εξελιχθεί προ όφελο των πολιτών. Κοιτάξτε, αυτή τη συζήτηση την κάνουμε μετά τις καλοκαιρινές ε, διακοπές και πράγματι έχετε δίκιο. Τα πράγματα δεν είναι άσπρα μαύρα. Υπάρχει και το γκρι, το γκρίζο, η φαιά ουσία. Πάμε στο 24. Αυτό αναβλήθηκε. Για το 25 δεν έχω τίποτα για τα διάφορα. 26. Ε, ανακοίνωση της επόμενης συνεδρίασης. 31 Αυγούστου. Και 31η... Όχι, με συγχωρείτε, 31 η οχι με 31 αυγουστου και 1η Σεπτεμβρίου. Τι... Ε, σας εύχομαι καλές διακοπές, ε, να ξεκουραστείτε. Ε, να γεμίσετε τις μπαταρίες σας για να επανέλθετε πιο ανανομένοι μετά τις ελληνές διακοπές. Ευχαριστούμε πολύ.